Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ο κύριος Μπούζεκ δεν μπορεί να προεδρεύσει σήμερα τη συνεδρίαση αυτή. Μου ζήτησε να το πράξω εξ ονοματός του. Να σας πω επίσης Ο εισηγητής ο κ. Γκρόμπασεκ δεν είναι παρόν, επειδή όμως είναι από την ομάδα ECR και εγώ επίσης, θα αναλάβω την χρονοθυρίδα του και λόγω της ε, υψηλής παρουσίας βουλευτών μάλλον θα πρέπει εγώ να παρουσιάσω το εγγραφό του. Η μερισσία διάταξη καταρχήν η οποία βρίσκεται εντός των φακέλων σας. Η πληροφόρηση σε σχέση με την επίσκεψη στην Ουασιγκτόνα έχει αναβληθεί μέχρι τις 7 Μαΐου. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν άλλα σχόλια μπορούμε να καλωσορίσουμε τους ομιλητές οι οποίοι έχουν δεχτεί και τους ευχαριστούμε τα μάλα να συμμετάσχουν στην ακρόασή μας αυτή. Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας πάντα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα ε, ανταγωνισμού στην αγορά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα. Πριν από 7 χρόνια περίπου ενεκρίθη το τρίτο ενεργειακό πακέτο με το στόχο να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό, χαμηλότερες τιμές και αποδεσμοποίηση της διανομής και παραγωγής ενέργειας. Έχει κυλήσει νερό κάτω από το αυλάκι έκτοτε αλλά δεν έχουμε ακόμα τέλειο ανταγωνισμό. Έχουμε προχωρήσει όμως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για την Ενεργειακή Ένωση και η Ήτρε αποφάσισε να συντάξει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και έχουμε αποφασίσει ότι ο κύριος Γκόρμπατσεκ θα είναι ο για το θέμα αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σχόλια που θα έκανε ο εισηγητής αν ήταν εδώ. Πολύ σύντομα και απλά. Τι θα μας έλεγε ο κ. Κρόμπατσεκ αν ήταν παρόν, εάν ερχόταν εγκαίρος ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της αγορά θα τόνιζε ενδεχομένω επίση το γεγονός ότι το μείγμα ενέργειας θα πρέπει φυσικά να εξακολουθεί να προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Και προσωπικά πιστεύω ότι βέβαια αυτές οι δύο προηγούμενες δηλώσεις μπορεί να αντιφάσκουν σε κάποιο βαθμό. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι το κόστος ενέργειας είναι κέριο για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και όλοι φυσικά έχουμε διαμαρτυρηθεί για την αποβιομηχάνηση πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να αναστρέψουμε αυτήν την τάση, αλλά αυτό απαιτεί φυσικά ένα πιο ανταγωνιστικό τίμημα ενέργειας, ενέργεια η οποία θα είναι σε ένα επίπεδο που θα είναι ανταγωνιστικό σε επίπεδο διεθνών τιμών. Για την οργάνωση της ακροασής μας θέλω να σας πληροφορήσω ότι έχουμε υπολογίσει τρεις ώρες και η ακρόαση θα είναι σε δύο τμήματα και θα υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις μετά από κάθε τμήμα. Ερωτήσεις και απαντήσεις θα κρατάνε περίπου 20 λεπτά και μετά ο πρόεδρος θα ζητήσει από τα μέλη της Επιτροπής μας να περιοριστούν σε δύο λεπτά σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις τους. Σας ευχαριστώ εάν τηρήσετε αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές ώστε να μπορέσουν και οι ομιλητές να απαντήσουν στα ερωτήματα στο τέλος. Το πρώτο πάνελ αφορά την μεγαλύτερη ολοκλήρωση για την αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, τις λύσεις που θα άρουν τα εμπόδια και το πώς θα πρέπει η Ενεργειακή Ένωση να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο το, στον πρώτο μας ομιλητή. Α, εδώ είσαστε. Μα όταν ξεκίνησα να μιλάω νόμιζα ότι δεν ήσασταν εδώ. Στον κύριο Ανδρέα Κουμπίλιας, ο οποίος είναι πρώην Πρωθυπουργός της Λιθουανίας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο και έχετε τώρα το λόγο για 10 λεπτά συναπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου δίδεται η δυνατότητα να πάρω το λόγο μπροστά σας. Θα σας μεταφέρω τις συγκεκριμένες εμπειρίες που έχουμε σωρεύσει στον τομέα της ενέργειας θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό ήταν για τη δική μας περίπτωση να ακολουθήσουμε την κοινή πολιτική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο μας βοήθησε αυτό να προχωρήσουμε και στα πλαίσια της απελευθέρωσης του συστήματος ενέργειας αλλά και της ολοκλήρωσής του με το ευρωπαϊκό σύστημα. Θα αναφερθώ στην προσωπική μου εμπειρία. Ήμουνα δύο φορές πρωθυπουργός της Λιθουανίας. Τελευταία φορά από το 8 μέχρι το 12. Το 2008 ήμουν τυχερός βέβαια που ε, ξεκίνησε στην ε, συγκεκριμένη συγκυρία η πρωθυπουργία μου αλλά είχαμε προβλήματα στον τομέα της ενέργειας γιατί μετά από 20 χρόνια πολιτικής ανεξαρτησίας ήμασταν εξαρτημένοι από τη Ρωσία στην ενέργεια. Πέραν τούτου και μετά από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε την υποχρέωση αναλάβει να κλείσουμε τα παλιά πυρηνικά ε, ε, ε, εργοστάσια στο τέλος του 2009 Επαναλαμβάνω ότι σε εκείνη τη φάση ήμασταν 100% εξαρτημένοι από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η εμπειρία μας λοιπόν είναι σαφής. Μόνο μέσω της χρήσης των μέσων της ευρωπαϊκής πολιτικής θα μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις αντιστάσεις της Gazprom ε, την προσπάθειά μας για ανεξαρτησία. Ε, ήδη από το 2009 αρχίσαμε να εφαρμόζουμε τα καινούργια μέτρα τα οποία είχαμε ε, πάρει. Πολλές μεταρρυθμίσεις και στον τομέα του φυσικού αερίου. Βασικός μας στόχος ήταν να αλλάξουμε την κατάσταση εξάρτησης του παρελθόντος. Έπρεπε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικέ πηγές φυσικού αερίου. Οι αντιστάσεις της Γκασπρόμ ήταν τεράστιες και σε πολιτικό και σε οικονομικό. Αλλά στη Βαλτική περιοχή ήμασταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες προχωρήσαμε σε τόσο μεγάλες αλλαγές. Η Γκάσπρομ προσπάθησε να σταματήσει αυτό που κάναμε. η Γκάσπρομ θέλησε να μην λειτουργήσουμε σαν αυτόνομες βαλτικές χώρες. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε πολλές αποφάσεις και κινήσεις της Γκάσπρομ ε, για πολιτικούς λόγους, αύξησε το κόστος του φυσικού αερίου ειδικά για τη χώρα μας σαν κύρωση, σαν τιμωρία. Όχι μόνο λοιπόν ήμασταν εξαρτημένοι κατά 100% από την Gazprom, αλλά λόγω και των πολιτικών αποφάσεων τις οποίες είχαμε λάβει, η Gazprom ήταν και κατά πλειοψηφίαν η της δικής μας εταιρείας. Κατανοήσαμε λοιπόν ότι όσο εφαρμόζαμε αυτό το ενεργειακό πακέτο, έπρεπε να προετοιμάζουμε και νέες δυνατότητες για εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Ήδη λοιπόν το 2010 ε, ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε ένα κέντρο αποθήκευσης ε, φυσικού αερίου. Μόνο μια τέτοια εγκατάσταση θα μπορούσε να μας δώσει κάποιο ποσοστό ανεξαρτησίας από την Gazprom και με αρκετά υψηλή ταχύτητα. Συναντήσαμε λοιπόν αντίσταση από την Gazprom, είμαστε και μικρή χώρα, 6 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά δεν σταματήσαμε τις μεταρρυθμίσεις μας, συνεχίσαμε Είχαμε ισχυρή πάντα βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Επίτροπο Έτιγκερ και την ομάδα του και γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες είχαμε προγραμματίσει. Χρησιμοποιήσαμε επίσης και τα μέσα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια. Το 2011 είδαμε ότι η Gazprom προσπαθούσε να μας σταματήσει να χρησιμοποιούμε αυτά τα οικονομικά και πολιτικά μέσα για μεταρρύθμιση. Προσφύγαμε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ζητήσαμε να διερευνήσει τις πρακτικές της Gazprom στην Λιθουανία και σε όλη την Κεντρική Ευρώπη. Θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή σύντομα. Το 12 ε, προσφύγαμε επίσης ε, και στη διαιτησία της Στοκόλμης και ζητήσαμε να μας αποζημιώσει με 8 ε, δις η Γκασπρόμ για την περίοδο 10 με 12 όταν οι τιμές της Γκασπρόμ δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικές. Και Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο, αυτό το οποίο έγινε τελικά είναι ότι εφαρμόσαμε το συγκεκριμένο πακέτο το οποίο ε, ήταν ε, πλέον λειτουργήσε το 2014. Ο τερματικός σταθμός αποθήκευσης τώρα πλέον ολοκληρώνεται και μπορούμε να εισάγουμε ποσότητες ε, θαλασσίως η Gazprom το 2014 αποφάσισε να μειώσει το κόστος του φυσικού αερίου κατά 20% και επίσης αποφάσισε η Gazprom να εγκαταλείψει πλήρως τις μετοχές τις οποίες είχε στην λιθουανική εταιρεία. Το συμπέρασμά μου λοιπόν είναι απλό. Χρησιμοποιώντας τα μέσα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας στον τομέα του αερίου, έχουμε εναλλακτικέ πηγές προμήθειας μέσω του τερματικού σταθμού NLG, εμείς τον χτίσαμε τον σταθμό αυτό με δικά μας χρήματα και μπορεί να καταστεί ε, κέντρο περιφερειακό και μάλιστα η Εσθονία θα αποθηκεύει και αυτή η ποσότητες φυσικού αερίου στο ε, τερματικό σταθμό των δικών μας. Στο μέλλον λοιπόν θα υπάρξει δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου σταθμού αυτού για πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, όχι μόνο για τις χώρες της Βαλτικής δηλαδή, αλλά και για την Πολωνία. Νομίζω ότι θα υπάρξει και η δυνατότητα κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου ανάμεσα στην Πολωνία και την Λιθουανία και μπορεί να έχουμε στο μέλλον μία σύνδεση και με την Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω πάρα πολύ σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη την πολιτική της ενέργειας, μια κοινή πολιτική και αποδίδει η πολιτική αυτή, ιδιαίτερα στην περιοχή μας. εφαρμόζοντας μια τέτοια πολιτική, πρώτον, είμαστε σε θέση να σπάσουμε την απομόνωσή μας την ενεργειακή, δεν είμαστε πλέον μια ενεργειακή νήσος, και νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ενεργειακής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Κουμπίλιους. Ε, επόμενος ομιλητής, επόμενη ομιλήτρια μάλλον η κυρία Κλάουντια Κέμφερντ είναι καθηγητής ε, ε, οικονομίας της ενέργειας και αηφορίας στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Hertie School of Governance του Βερολίνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και με μεγάλη χαρά εμφανίζομαι ενώπιόν σας. Έχω ενημέρωση για το σύνολο των προκλήσεων για την εσωτερική αγορά ενέργειας με ιδιαίτερη στόχευση στην αγορά ενέργειας και στην κοινότητα ενέργειας, την Ένωση Ενέργειας. Ποιες είναι οι προκλήσεις. η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να αποτελέσει όθηση για μια αλλαγή στην ενέργεια. Ποιοι είναι οι στόχοι. Για πρώτη φορά έχουμε 80% στόχο μείωσης των εκπομπών από το επίπεδο της Ένωσης. Για να φτάσουμε τον στόχο αυτό πρέπει να μπούμε και στον τομέα της ενέργειας και σε άλλους τομείς. Υπάρχει η πρόκληση τώρα να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος ε, για το 2050. Αν δούμε το 2020 βλέπουμε στη διαφάνεια αυτή ότι υπάρχει διαφορετική εξέλιξη ανά χώρα μέλος. Εξετάστε την διαφάνεια και θα δείτε ότι υπάρχει σημαντική μείωση των εκπομπών σε ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Δεν βλέπετε τις διαφάνειες. δεν φαίνονται από ό,τι φαίνεται διαφάνειες. Πάντως θα δείτε και αυξήσεις σε ορισμένες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι η πρόκληση για το 2020, αλλά και για να επιτευχθεί ο στόχος του 2050 θα είναι σημαντικό να ληφθούν και άλλα μέτρα και να προβλεφθούν και άλλα εργαλεία για να επιτευχθεί ο στόχος. Αν δούμε τώρα τα όργανα που έχουμε, βλέπετε μια τιμή του τόνου του διοξιδίου του άνθρωπος που είναι υπερβολικά χαμηλή και αν μείνουμε εκεί πολύ δύσκολα θα φτάσουμε και μακροπρόθεσμα, δηλαδή 2050, στον στόχο. Ε, βρισκόμαστε στα 7 ευρώ τον τόνο για την ώρα και για να είναι σημαντική η επίπτωση θα πρέπει η τιμή να είναι πολύ ακριβότερη, πολύ υψηλότερη. Πάντως δεν έχουμε στόχο μόνο της μείωσης των εκπομπών, έχουμε και στόχο για τις ανανόσιμες ενέργειες που έχουμε σχεδόν επιτύχει, θα έχουμε σχεδόν φτάσει τον στόχο. Η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να αποτελεί βέβαια πρόκληση αλλά και ευκαιρία για πιο μακροπρόθεσμους στόχους για τις ανανεώσιμες ενέργειες και πρέπει να επιτύχουμε τους επιμέρους στόχους και εδώ βλέπετε και εδώ την διαφάνεια που αναφέρει τις διάφορες χώρες που καλά τα πάνε λίγο πολύ αλλά όπως είπα είναι και μακροπρόθεσμος ο στόχος. Τώρα αν εξετάσουμε τα όργανα που διαθέτουμε. Πρέπει να υπάρχει την αρμόνιση των κανόνων και μέτρων. Βλέπετε ένα σύστημα ε, τέλους τροφοδοσίας και πρημοδότησης και βέβαια και ποσοστώσεις. Βλέπουμε και τάσεις που προέρχονται τώρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξουν περισσότεροι διαγωνισμοί, αυτό γίνεται δηλαδή η προκήρυξη διαγωνισμών, αυτό γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει σε πολλές, γίνεται στη Γερμανία για παράδειγμα, αλλά εξακολουθεί η συζήτηση αν θα πρέπει να υπάρξει αυτό το tendering system. Τώρα για τα ορυκτά καύσιμα βλέπετε ότι και εδώ υπάρχουν πολλές επιδοτήσεις για ανανεώσιμες ενέργειες αλλά και για τα ορυκτά καύσιμα θα δείτε και τη σύγκριση ότι τα ορυκτά καύσιμα λαμβάνουν επιδοτήσεις περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια με διαφορές ανάμεσα στις χώρες, αλλά και ανανεώσιμες ενέργειες έχουν ένα σύστημα κινήτρων. Το ερώτημα είναι βέβαια εάν θα πρέπει και αυτό να εναρμονιστεί. Μου ζητήσατε να σας μιλήσω και για τις ε, επενδυτικές στρατηγικές που απαιτούνται. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το σενάριο που θα εξετάσει κανείς. Αν εξετάσουμε ένα καθαρό σενάριο πράσινης μετάβασης ή αν θα είναι ταχύ ή λιγότερο ταχύ, βεβαίως οι νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, βελτίωση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, επίσης η προσπάθεια να μειωθούν εκπομπές με χρήση διαφόρων τεχνολογιών, αλλά και για την συζήτηση είναι σημαντικό αυτό τώρα για τις υποδομές για να βελτιωθεί το όλο σύστημα όχι μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και για το φυσικό αέριο. Ακούσαμε ήδη σχετικά με το φυσικό αέριο που είναι κρίσιμο βέβαια διότι η εξάρτηση από τη Ρωσία εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή. Βλέπετε όπως ακούσαμε και λίγο πριν σημαντική εξάρτηση από τη Ρωσία για πολλές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και για τις βαλτικές χώρες. Το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτηση αυτή και τι μπορούμε να πράξουμε σχετικά. Εμείς έχουμε κάνει εδώ μια μελέτη του ε, Γερμανικού Ινστιτούτου DIV που δείχνει ότι μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτηση και να βελτιώσουμε την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. Αυτό είναι κρίσιμο βεβαίως για να βελτιωθεί η ασφάλεια θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία και μπορεί να μειωθεί κιόλας με μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εισαγωγών αερίου από τη διεθνή αγορά. Διότι υπάρχει επαρκές αέριο στην ε, ε, διεθνή αγορά και μάλιστα το υγροποιημένο φυσικό αέριο παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να αυξηθεί ε, η ποσόστοσή του. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν. Έχουμε δει επίσης πολλούς τερματικούς εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βεβαίως έχουμε τώρα και στη Γερμανία. Για να μειωθούν οι εισαγωγές από τη Ρωσία και για να διαφοροποιηθούν οι εισαγωγές. Τώρα, κάναμε και μια μελέτη που βλέπετε εδώ για την κυριότητα από πλευράς Gazprom των αγωγών, του δικτύου δηλαδή διανομής, βλέπουμε σε διάφορους αγωγούς την κυριότητα αυτή όπως το Nord Stream και σε άλλους, αλλά και σε επιλογές αποθήκευσης. Επίσης η Gazprom διαθέτει και δίκτυα ή τουλάχιστον ποσοστά σε δίκτυα διανομής του αερίου και στη Γερμανία αλλά και στη Σερβία και αλλού. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί η διαφοροποίηση και των εισαγωγών αλλά να εξεταστεί προσεκτικά και η κυριότητα ποσοστών στα δίκτυα της Gazprom. Αυτά είναι βέβαια και μέσα σε δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς. Επίσης σημαντική είναι η υποδομή για την ενέργεια για να βελτιωθεί η Ένωση Ενέργειας. Βεβαίω τα αποτελέσματα διαφέρουν αναμελέτη. Εμείς έχουμε κάνει εδώ και εξομοιώσεις και βλέπετε τα αποτελέσματα. Υπάρχει αναγκαιότητα επένδυσης στα δίκτυα, αλλά και όχι μόνο. Γιατί είναι σημαντικό για να βελτιωθεί η ασφάλεια προμήθειας ενέργειας και για να βελτιωθεί και το υφιστάμενο σύστημα πρέπει Βεβαίω εξαρτάται πάντοτε από τη μελέτη που κοιτάζει κανεί, αλλά φαίνεται να είναι απαραίτητο μέχρι το 2030 να επενδυθούν 30 δισεκατομμύρια. Σημαντικό αυτό για να αποφευθούν και τα σημεία εχμής και όχι μόνο στο ηλεκτροδοτικό σύστημα. Πάλι και για το φυσικό αέριο κάναμε και εδώ μια μελέτη και για άλλα και πρέπει να επενδύσουμε και σε υποδομές διανομής του φυσικού αερίου. Βεβαίως εκεί σημειώνονται διαφορετικές διαφορετικά σημεία εχμής και στην Νότια Ευρώπη και πρέπει και εκεί να γίνει προσπάθεια βελτίωσης και να βελτιστοποιηθούν τα συστήματα διανομής του φυσικού αερίου και να βελτιωθούν και οι ροές αποδυσμάς δηλαδή προς Ανατολάς. Επίσης σημαντική είναι η Νορβηγία από την άποψη αυτή και για τη βελτίωση βέβαια του συστήματος έρχομαι στο τέλος σιγά σιγά, η Ενεργειακή Ένωση προσφέρει πολλές προκλήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες είναι όχι μόνο ότι πρέπει να υπάρξει μικρότερη εξάρτηση για τις προμήθειες ενέργειας από άλλες περιοχές του κόσμου όπως από τη Ρωσία και την αγορά αερίου της, αλλά να δοθεί και μια ευκαιρία επίτευξης πιο μακροπρόθεσμων στόχων για να επιτεθεί και να, να και να επιτεθεί η μετάβαση σε ε, άλλες ενέργειες. Και τι γίνεται βέβαια και με τον στόχο των ανανεώσιμων ενέργειων, ε, ε, αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, καθώς και μείωση των εκπομπών. Και εδώ έχουμε βέβαια και, τις, και τους στόχους 2030. Από στην πλευρά των ανανεωσίμων χρειαζόμαστε συστήματα στήριξης χαμηλού κινδύνου απαραίτητο εδώ να αναλυφθεί ταχύως ενέργεια γιατί βελτιώνει αυτό βέβαια την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας και όσο βελτιώνεται η ασφάλεια προμήθειας ενέργειας τόσο λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιούμε εν τέλει άρα είναι και πιο αποδοτική η χρήση της και πάλι αυτή με τη σειρά της ε, ανεβάζει την ασφάλεια ενέργειας. Για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακο επίση χρειάζονται κάποια μέτρα όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά βέβαια και εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων. Εν τέλει το συμπέρασμα μου είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε ένα όραμα για την Ενεργειακή Ένωση, βλέποντας ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, διότι η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να αποτελέσει την όθηση για την μετάβαση στην ενέργεια για διάφορες επιμέρους χώρες, μπορεί να επιφέρει και καινοτομία, θα πρέπει να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, να μειώσει το κόστος των ανανοσίμων ενεργειών και να εξασφαλίσει ότι στο μέλλον θα είναι φθηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος κύριε Κέμφερτ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ε, υποβολή ερωτήσεων. Επειδή φορώ και την κασκέτα του συντονιστή του ECR, της συντηρητικής και μεταρρυθμιστικής ομάδας, θέλω να θέσω το πρώτο ερώτημα, που είναι κάπως ακαδημαϊκού χαρακτήρα ερώτημα και για τους δυο Λέμε από τη μία πλευρά ότι θα θέλαμε να είχαμε εθνική λήψη αποφάσεων για το μείγμα ενέργειας. Είναι ένας τεθειμένος στόχος. Ο άλλος στόχος όμως είναι να εξασφαλίσουμε μια πραγματική κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Το ερώτημά μου είναι συνάδουν αυτοί οι δύο στόχοι ή συγκρούονται μεταξύ τους. <clears throat> Το επόμενο ερώτημα, ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, παρουσιαστές μας. Νομίζω ότι ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια του ΕΛΚ να προχωρήσουμε προ μια ενεργειακή ένωση και ιδίως τονίζοντας τη σημασία του να έχουμε σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και έτσι να αντισταθμίσουμε την ανάγκη να εξαρτώμαστε πάντα από τη Ρωσία. Από πρακτική όμως έποψη, πόσους θερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου θα πρέπει να έχουμε στην Ευρώπη για κάθε χώρα και πώς θα συνδεθούν με το δίκτυο ώστε να έχουμε την μέγιστη ε, διασύνδεση. Για το θέμα της ανανεώσιμης ενέργειας τώρα. Μήπως υπάρχει κάποια δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια συνέργεια μεταξύ τερματικών σταθμών LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, και ενεργειακών ε, αγροκτημάτων όπως λέγονται, δηλαδή εξωχώριων, μάλλον θαλασσίων σταθμών ε, αιωλικής ενέργειας. Μήπως μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα αυτοί οι δύο τρόποι παραγωγής, αυτοί οι δύο, ε, αυτές οι δύο υποδομές ενέργειας. Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε και η οικονομία κλίμακος με το να έχουμε διαφορετικούς τομείς ενέργειας να συνεργάζονται μεταξύ τους και να έχουμε έτσι μία κοινή υποδομή και όχι μονάχα να λειτουργούν απομονωμένα και διάσπαρτα. Ακολουθεί το ερώτημα της κυρίας Τόγια από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Αναφέρομαι στην κυρία Κέμφερτ που έκανε το, τη δεύτερη παρουσίαση. Εντάξει. Έλεγα ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω για να καταλάβουμε λιγάκι καλύτερα ποια είναι τα θέματα αυτά. Γι' αυτό κάνω δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, για τα 10 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων που δίδονται τώρα σε γενικό ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την χρήση των ε, συμβατικών καυσίμων, των ορυκτών καυσίμων. Μήπως μπορούμε να ξέρουμε κάτι περισσότερο για την κατανομή αυτών των επιδοτήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για να καταλάβουμε καλύτερα σε τι συμπεράσματα φτάνει η μελέτη σας. Και κατά την δική σας άποψη θα ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα, ίσως μπορεί να το δει κανεί και από τα στοιχεία σας, αλλά επειδή είναι κάπως δύσκολο να το βρω από την διαφάνειά σας, τι <coughs> εξασφαλίζει αυτό ή δεν εξασφαλίζει σε επίπεδο θεμητού ανταγωνισμού στα επίπεδα ενέργειας. Πώς λοιπόν μπορείτε να εκτιμήσετε τις συνέπειες αυτής, αυτών των επιδοτήσεων. Το δεύτερο ερώτημα είναι πολύ πιο σύντομο. Έχει να κάνει με τις προβλέψεις για επενδύσεις στον, εργασί, στον ενεργειακό τομέα. Από ό,τι κατάλαβα, η μελέτη του DIV e του Βερολίνου μιλάει για 30 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας, μάλλον φτάνοντας μέχρι το 2030 σε επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Οι τα διαφορετικά αυτά σενάρια έχουν να κάνουν με διαφορετικές ε, προβλέψεις και βλέπω εκεί τον πίνακα που αναφέρεται σε προβλέψεις για επενδύσεις για την ε, ηλεκτροδότηση. Έρχονται αυτά από το δικό σας ίδρυμα Υπάρχουν τα 30 δισεκατομμύρια που αναφέρει το Ίδρυμα το ΔΕΙΒΕ. Υπάρχουν άλλες μελέτες και μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι μελέτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλικιώτης έχει το επόμενο ερώτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Η ανάγκη ενίσχυση τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αερίου αποτελεί σήμερα μια βασική προπόθεση για να έρθει η ενεργειακή απομόνωση, στην οποία βρίσκονται πολλά κράτη και περιοχέ τη Ευρώπη. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ο μιλητή, ο κύριο ε, ε, Κουπίλιου, ε, ότι η Λιθουανία ξεπέρασε τα προβλήματα, αλλά την ίδια ώρα γνωρίζουμε ότι χώρε, κράτη-μέλη τη Ανατολική Ευρώπη και της Μεσογείου και περιοχές είναι απομονωμένες από την πρόσβαση σε φυσικό αέριο αλλά και από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Όπω βασική προπόθεση είναι η ενίσχυση αυτή τη αγορά ε, για την ενεργειακή ασφάλεια τη Ένωση, στην οποία σήμερα πάρα πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι σημαντικό να υπάρχουν οι απαραίτητε υποδομέ, ώστε να επιτύχουμε μια πλήρω ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη είναι στην εσωτερική αγορά ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αερίου, διασφαλίζοντα πρώτιστα την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών ε, σε ευθυνή ενέργεια ε, ή ακόμα και έναν υποστηρικτικό πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίων χαμηλού, χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, και οι διασυνδέσει με ρίχτη αγωγού και μεταφορικού δρόμου μπορεί να ενδυναμώσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συζήτητες. Πρώτα, πώς θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των στόχων τα, η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρουμε στη Μεσόγειο διότι η Μεσόγειο σήμερα υπάρχουν κράτη-μέλη και περιοχές που είναι απομονωμένα και από την ε, παροχή φυσικού αερίου αλλά και από την ενεργειακά δίκτυα και ε, πώς ε, βλέπουν την προοπτική δημιουργίας ε, σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Νότια Ευρώπη και αναφέρομαι σε και σταθμούς από υγροποίησης αλλά ενδεχομένω σε σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου. Γιατί εκεί υπάρχει πρόσβαση σε αγορές φυσικού αερίου και από την περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και της ε, ε, Βόρειος Αφρικής. Άρα ε, θα ήθελα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα και αναφέρομαι σε αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά για να υλοποιήσουμε του στόχου τη άρση τη απομόνωσης και τη ενεργειακή ασφάλεια ιδιαίτερα τη Νότια Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Okay, Σας ευχαριστώ, αλλά να τηρήσουμε όλοι τα δύο λεπτά παρακαλώ. Από την EFTD, ο κ. Θα είμαι πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με χαρά που αρχίζουν να μιλούν για λιγότερη χρήση ορυκτών καυσίμων. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται πράγματι να εξεταστεί το θέμα, ιδίως γιατί η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να έχει ως στόχο να μειώσει την εξάρτηση και θα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος τελικά ωφελείται από τις επενδύσεις και για λόγους δηλαδή διατήρηση του ανταγωνισμού. Και να υπάρξει βέβαια και αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Ε, για μένα μπαίνει το ερώτημα μήπως δεν θα είναι πιο δίκαιο να χρησιμοποιηθούν οι επενδύσεις αυτές ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια που αυξάνεται σε πολλές ε, χώρες μέλη και κυρίως αυτές που χτύπησε πιο πολύ, στις χώρες αυτές που χτύπησε πιο πολύ η κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πατσίτης έχει το επόμενο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εκπρόσωπο της Λιθουανίας που αντιμετώπισε την κρίση, την ενεργειακή κατά πρόσωπο και χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Ο κ. Κουμπίλιος αντιμετώπισε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Σήμερα έχουμε αυτού τους στόχους ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσουμε τις εκπομπές αριών του θερμοκηπίου, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους ανανεώσιμους πόρους, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε ένα πρόβλημα όμως έλλειψης αλληλεγγύης. Πιστεύουν οι ομιλητές μας ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή να σκεφτούμε περισσότερο και πιο σοβαρά στη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να καταδείξουμε στα άλλα κράτη ότι αυτό θα ήταν μια πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν μια πολύ χρήσιμη απόφαση. Για να εξηγηθώ καλύτερα. Η Λιθουανία είχε μια σύνδεση σε επίπεδο φυσικού αερίου με την Πολωνία. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε αυτήν την σύνδεση φυσικού αερίου, γιατί είχαμε απλώς και μόνο μία σύνδεση ε, σε επίπεδο ηλεκτροδότησης και είμαστε αναγκασμένοι να παίρνουμε φυσικό αέριο από τη Γερμανία. Τονίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αυτό το σχέδιο, αλλά θέλουμε να γίνει μια χρηματοδότηση σε επίπεδο γενικότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μονάχα από τις βαλτικές χώρες και την Πολωνία. Εδώ τίθεται το θέμα της αλληλεγγύης. Θα πρέπει ίσως να καταλάβουμε ποιες είναι που έχουν αναλάβει οι χώρες μέλη για να εξασφαλίσουν μια πραγματική ενεργειακή ένωση. Θα πρέπει εκεί το κάθε κράτος μέλος να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο και εγώ πιστεύω ότι η δημιουργία μιας ενεργειακής αγοράς σε τελική ανάλυση θα αποβεί προς όφελος όλων των κρατών μελών. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπένσεν. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα προς την Κλαβδία Κέμφερτ. Εγώ ανησυχώ λιγάκι όταν βλέπω το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του δικτύου μας στην Ευρώπη έχει ιδιοκτήτες ξένους, ιδίως την Gazprom, η οποία ελέγχει και είναι ιδιοκτήτης πολλών δικτύων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήματα. Θα σας δώσω κύριε Κουμπίλιους πρώτα το λόγο σε εσά και μετά στην κυρία Κέμφερ. Πέντε λεπτά ο καθένας για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαν πολλά ερωτήματα που κάποια επικαλυπτόντουσαν κάπως μεταξύ των διαφόρων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα είναι το πώς, το πώς μπορεί να συνδυάζει κανείς τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. στα πλαίσια της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας. Αυτό το οποίο έχουμε εμεί αντιμετωπίσει υπό το φως αυτού θα ζητήσω περισσότερες εξουσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να προχωρήσει σε περισσότερα προγράμματα υποδομών με ισχυρότερη περιφερειακή διάσταση. Στην περίπτωσή μας, μιας και είμαστε απομονωμένοι θα έλεγα, έπρεπε να προχωρήσουμε πολλά περιφερειακά προγράμματα όπως διασύνδεση με το δίκτυο της Σουηδίας ε, ηλεκτρικό ε, εισαγωγή επίσης ε, ποσοτήτων φυσικού αερίου από τη Φιλανδία, από την Πολωνία κτλ. Οι εμπειρίες μας λοιπόν είναι συγκεκριμένες και απλές. Απαιτείται και κάποιος πατριωτισμός αν θέλετε, τοπικισμός να το πω αλλιώς. Είναι ένα μέσο ισχυρό για την αντιμετώπιση της δυσκολίας. Όταν εμείς ξεκινήσαμε τις μεταρρυθμίσεις στο φυσικό αέριο, ξέραμε ότι οι Ρώσοι θα ήταν πολύ εκνευρισμένοι. και ότι αν καθυστερούσαμε με την κατασκευή της, του τερματικού αποθήκευσης θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με τους Ρώσους. Και γι' αυτό είπαμε ότι ε, το να υπάρξει ένας περιφερειακός θεματικός σταθμός για τις τρεις χώρες θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο. Για να συμφωνήσουμε για τη διασύνδεση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος απαιτήθηκαν πάρα πολλά χρόνια όπως ε, ηλεκτρισμός από τη Σουηδία, σύνδεση με το Σουηδικό δίκτυο, εν πάση περιπτώσει για τη Λετωνία και τη Λιθουανία, ήταν χρονοβόρες οι διαδικασίες. Αυτό λοιπόν ε, το πρόγραμμα για περιφερειακό τερματικό είναι κάτι το οποίο θα καθυστερούσε πολύ. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί αλλιώς ε, τότε πράγματι θα μας είχε πνίξει η Gazprom αν δεν το είχαμε κάνει, αν δεν είχαμε κάνει την επιλογή αυτή. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα τερματικό με καλή χωρετικότητα που λειτουργεί με ασφάλεια. Θα ήταν καλύτερα όμως να είχαμε ένα διαφορετικό μέσο στη διάθεσή μας Αν είχαμε την Επιτροπή να μας καθοδηγεί βέβαια για περιφερειακής διάστασης έργα, προφανώς θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε ανάγκες μερικές φορές έναν ανώτερο διαιτητή για να μας καθοδηγεί και να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Αυτή λοιπόν ήταν η πρόκληση την οποία αντιμετωπίσαμε να ξεφύγουμε από το ρωσικό εναγκαλισμό αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσουμε και σε μια ευρύτερη περιφερειακή ε, διάσταση σε συνεργασία με την υπηρετική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία να προσπαθήσουμε να δούμε τι χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, να ξεπεράσουμε τους κόπελους των διαπραγματεύσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτείται να έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες και στα πλαίσια της οικοδόμησης δικτύων υποδομών για το σύνολο της Ένωσης. Λοιπόν, αυτές είναι οι απαντήσεις μου για το πώς εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε στις ε, υποδομές. Εγώ είμαι υπέρ των θερματικών φυσικού αερίου. Θα μπουν σύντομα και οι Αμερικανοί στην αγορά, οι τιμές θα κατέβουν μάλλον περισσότερο Ας μην είμαστε αυστηρά εξαρτημένοι από τις μεταφορές μέσω αγωγών. Μέσω της δημιουργίας αυτών των τερματικών ακόμα και σε άλλες περιοχές μπορεί να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας των προμηθείων. Τώρα για την αλληλεγγύη Νομίζω για να υπάρχει αλληλεγγύη πρέπει να δώσουμε δύναμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη για τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εδώ απαιτείται πολύ ισχυρότερη πολιτική παρέμβαση από πλευράς της Ένωσης και θα κλείσω λέγοντας ότι υπάρχουν περισσότερες ανάγκες για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας να υπάρξουν περισσότερο εναρμονισμένες, ενιοποιημένες ρυθμίσεις στις διάφορες χώρες όταν έχουμε να κάνουμε με μονοπόλια εθνικά όπως κάνουμε σαν παράδειγμα στην Τραπεζική Ένωση και στην ενέργεια να κρατήσουμε μια ενιαία στάση και στα πλαίσια της χορήγησης επιδοτήσεων. Ευχαριστώ κύριε Κέμφαρτ και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα που θέσατε. Σε πέντε λεπτά δεν μπορώ να απαντήσω στα λεπτομεριακά ερωτήματα για τα ίδια ορυκτών καυσίμων που πρέπει να προκρίνουμε, για τις διαφορές που υπάρχουν σε επίπεδο υποδομών, επενδύσεων. Θα μπορούσαμε να σας στείλουμε πιο λεπτομεριακά αριθμητικά στοιχεία και τις ε, μεμονωμένες μελέτες που έχουμε κάνει ιδίως σε ό,τι αφορά τις ε, επιδοτήσεις για συμβατικά ορυκτά καύσιμα, για τις επιδοτήσεις για τον άνθρακα, παραγωγικά στη Γερμανία, αλλά και διάφορες εξαιρέσεις από φορολογία. Πες περιπτώσει νομίζω ότι το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και για τις επενδύσεις σε δίκτυα διανομής. Έχουμε διαφορετικές εδώ απόψεις σε σχέση με το τι είδους υποδομές είναι απαραίτητες. Βλέπουμε να υπάρχουν σημεία συμφόρηση μεταξύ μερικών χωρών που θα έπρεπε να αρθούν για να βελτιωθεί το σύστημα. Και εδώ το θέμα τη αλληλεγγύη. είναι εξόχω σημαντικό γιατί η αλληλεγγύη θα πρέπει να παίξει και κάποιο ρόλο όταν δούμε το σύστημα των αγωγών φυσικού αερίου, παραδείγματο χάρη στι νότιε και ανατολικέ χώρε, εκεί πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να μπορούμε να έχουμε και ανάστροφη ροή για να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ να έχουν ενεργειακή ασφάλεια εκεί που είναι δύσκολο να πάρει κάνει το φυσικό αέριο στη διεθνή αγορά. Το ίδιο για τη μελέτη σε σχέση με την Gazprom. Μπορούμε να σα στείλουμε και αυτή, γιατί έχουμε εκεί αποτυπώσει τις ε, ανησυχίες μας για τα θέματα ασφάλειας τροφοδοσίας ε, σε ενέργεια. Το θέμα λοιπόν αυτό της ασφάλεια τροφοδοσίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί υπάρχει μεγάλη ε, παρουσία της Gazprom όχι μόνο στην ιδιοκτησία δικτύων αλλά και στους σταθμούς αποθήκευσης. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου όχι μόνο σε χώρες ε, κεντρικές όπως η Γερμανία αλλά και αλλού είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφοροποίηση και υπάρχει πραγματικά αρκετό υγροποιημένο αέριο στη διεθνή αγορά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Απλώς κάποιοι τερματικοί σταθμοί δεν, δεν ε, έχουν τύχει πλήρους ε, εκμετάλλευσης, αλλά από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να του χρησιμοποιήσουμε θα μειωθεί και η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αλληλεγγύης. Μέχρι ότου μπορούμε να φτάσουμε την Ενεργειακή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια αλληλεγγύη. Για το θέμα της εναρμόνισης, για το πόσο εναρμονισμένο θα πρέπει να είναι το σύστημα σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, Αυτό φυσικά παραμένει στα χέρια των εθνικών αρχών για το ενεργειακό μείγμα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε είναι να εναρμονίσουμε το γενικό πλαίσιο επιδοτήσεων, να απαραίτητο να έχουμε κοινού στόχου, όχι μονάχα για τη βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση, τι ανανεώσιμε ενέργειε, αλλά και κοινού στόχου για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και αυτό δεν αφορά μονάχα τι βαλτικέ χώρε, αλλά και τι χώρε τη ε, νότια-ανατολικής Ευρώπη που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες αν δεν βελτιώσουμε το σύστημα των αγωγών φυσικού αερίου και δεν γίνει πιο αποτελεσματικό θα είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε τα πρότυπα ενεργειακής <clears throat> ασφάλειας τροφοδοσίας που θέλουμε να έχουμε για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο θα παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον για την Ενεργειακή Ένωση. Δεν το χρειαζόμαστε μονάχα για την ενεργειακή μετάβαση αλλά θα μπορούσαν να συνδυαστούν σταθμοί παραγωγής με φυσικό αέριο με σταθμούς ανανεώσιμης ενέργειας που μας δίνει αυτό μεγαλύτερη ε, ευελιξία και επίσης και για την αγορά ενέργειας κινητικότητας όπου μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο το φυσικό αέριο. Έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία της Ενεργειακής Ένωσης, θα πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά και να καταλήξουμε σε ένα κοινό πλαίσιο που να καλύψει όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και, τον κύριο Κουμπίλιους για την παρουσίασή του επίσης. Τελείωσε το πρώτο τμήμα της ακρόασής μας. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους άλλους ομιλητές που βρίσκονται στο δεύτερο πάνελ να έρθουν <clears throat> εδώ στα προεδρικά θεωρία. Παρακαλώ, ελάτε. Και ενδιαμέσως σας ανακοινώνω τον τίτλο του δεύτερου πάνελ. Μιλάμε για το λόγο της ε, εγχώριας παραγωγής ενέργειας, εξασφάλισης των διασυνδέσεων για την αγορά από ανανεώσιμες ενέργειες ηλεκτρισμού και τα θέματα της, μειώση, της μείωσης των ε, εκπομπών. Ξεκινώ με τον κύριο Λούις Ατιένδα, ο οποίος είναι ε, επικεφαλής του, της σχολής ε, του, Duisburg, και ήταν διευθύνων σύμβουλος της ε, RD e Electrica στην Ισπανία που είναι ένας, ε, φορέ, ένας, ένας φορέας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριε Ατιένσα, έχετε το λόγο για 10 ολόκληρα λεπτά περίπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι κοινοβουλευτικοί, Ευχαριστώ και το, την Επιτροπή σας που μου δίνει την ευκαιρία να συμμεριστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις που προέρχονται από την εμπειρία μας σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα <clears throat> σε ό,τι αφορά τον τομέα της ηλεκτροδότησης. Το πρώτο που θέλω να αναφέρω είναι το γεγονός ότι οι φορείς αυτής της μετάβασης δεν είναι αυτό που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πριν από 15 20 χρόνια, δηλαδή ότι θα ήταν αποτέλεσμα της εξάντλησης των φυσικών πόρων, αλλά περισσότερο από την πολιτική για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και είναι επίσης αποτέλεσμα της τεχνολογικής βελτίωσης. Πρόκειται για την ορίμανση των τεχνολογιών χωρίς ε, χρήση διοξιδίου του άνθρακος, φωτοβολταϊκά και ολική ενέργεια, είναι η βελτίωση των ε, τεχνολογιών για την αποθήκευση ενέργειας, για την αυτόματη διαχείριση των, ε, της κατανάλωσης και επίσης για την πολιτική κατάσταση κλιματικής αλλαγής που γίνεται τώρα ένα βασικό συστατικό στοιχείο των αποφάσεων που παίρνουν οι καταναλωτές και οι εθνικές αρχές. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θέτει το ηλεκτρικό σύστημα, σύστημα ηλεκτροδότησης, στο κέντρο της πολιτικής απεξάρτησης από τον άνθρωπο για την ενέργεια. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι αυτή η τεχνολογική μεταλλαγή, ουσιαστικά η ορίμανση ορισμένων τεχνολογιών που οδηγούν σε οικονομία, σε χαμηλού επίπεδου οικονομίας κλίμακος, η ανάπτυξη των τεχνολογιών διαχείρισης της ε, ζήτησης θα οδηγήσουν σε μια μετακίνηση, σε μια σημαντική μετακίνηση του κέντρου βάρους του ηλεκτρικού συστήματος από μια συγκεντρωτική παραγωγή προ μια παραγωγή που είναι πολύ πιο κοντά προ του καταναλωτέ. Αυτό σημαίνει αποκέντρωση και δημοκρατικοποίηση της ενεργειακή τροφοδοσίας στο βαθμό που μπορεί να εξασφαλίσει μια πιο ενεργή, ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών οι οποίοι είναι και εν μέρη παραγωγή ενέργειας. Αυτή λοιπόν η τροποποίηση του μείγματος ενεργειών και η μετακίνηση προς μια αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας σημαίνει και σημαντικές τεχνικές αφενός προκλήσεις και επίσης προκλήσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά το σύστημα ηλεκτροδότησης που προφανώς έχουν επιπτώσεις και για την αγορά ε, ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ενεργειακή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προκλήσεις προκύπτουν από την ανάγκη να διαχειριστούμε ένα σύστημα ηλεκτροδότησης όπου υπάρχει πολύ μεγάλο τμήμα διαλύπουσας παραγωγής ενέργειας, μεταβλητής δηλαδή ε, παραγωγής ενέργειας που έχει και μεγάλη γεωγραφική διασπορά και αποκέντρωση. Αυτό αφορά κυρίως την αιωλική ενέργεια. Και επίσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η από την δομή των δικτύων όπως στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών ή της ε, συμπαραγωγής ενέργειας. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του συστήματος εν ώψη της διακύμανσης της ζήτησης και να εξασφαλίσουμε ότι θα μεταφέρεται η ενέργεια εποφελώς από τις περιοχές παραγωγής, περιοχές κατανάλωσης. Οι απαντήσεις σε αυτό θα πρέπει να προκύψουν καταρχήν από την εξέλιξη των συστημάτων έλεγχου και παρακολούθησης στην Ισπανία έχουμε προωθήσει τη δημιουργία του ΘΕΚΡΕ που είναι ένα κέντρο ελέγχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό μπόρεσε να διαχειριστεί την πολύ μεγάλη μεταβλητότητα της παροχής αιωλικής ενέργειας. Θα πρέπει να καταλάβετε το ισπανικό σύστημα από το υψηλότερο ως το χαμηλότερο επίπεδο έχει διαφορά 17.000 ε, ΜΒ για τα για την αιωλική ενέργεια, αλλά είναι μόνο 1.400 ΜΒ η ικανότητα διασύνδεση με το ευρωπαϊκό σύστημα. Επομένω, θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου τη χρήση των ανανεώσιμων ενεργειών και έχουμε ήδη προχωρήσει σημαντικά στην συμβολή που μπορεί να γίνει από τους μηχανισμούς αυτόματου ελέγχου του συστήματος αλλά θα πρέπει να, απο, να δημιουργήσουμε και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, <clears throat> όπως είναι η άντληση ύδατος ως ένα αντιστρεπτό σύστημα αποθήκευσης και επίσης τα συστήματα ε, αποθήκευσης με συμπίεση ε, αερίου ή με ηλεκτροσυσσωρευτές, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε θα υπάρξει μία ε, προσαρμογή της προσφοράς τη ζήτηση μέσα στο σύστημα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στις διασυνδέσεις για τον ηλεκτρικό ε, τομέα. Αν έχουμε ένα σύστημα απεξαρτημένο από τον άνθρακα ε, θα απαιτεί πολύ μεγάλη ικανότητα του δικτύου για να μπορέσει να διαχειρίζεται σωστά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τις περιοχές ε, Παραγωγή στι περιοχές κατανάλωση. Χρειάζεται ένα ιδιαίτερα ευφυές σύστημα για να μπορεί να ελέγχει την μεταβλητότητα και την ανάγκη τροποποίηση τη ζήτηση μεταξύ των χωρών μελών, ώστε όχι μονάχα να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα μέσω των διασυνδέσεων για τους καταναλωτές, αλλά συγχρόνως εξασφαλίζεται και η τεχνική ευρωστία του συστήματος και μας επιτρέπει το ηλεκτρικό αυτό σύστημα, το οποίο έχει την καλύτερη δυνατή διασύνδεση να μπορεί να αντιμετωπίζει την μεταβλητότητα της παραγωγής ηλεκτρισμού. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι οι συνέπειες που πρέπει να προκύψουν για τους ρυθμιστές και τον κανονιστικό τομέα. Το δεκαετία του 1990 το ηλεκτρικό μας σύστημα δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα τελείως διαφορετικό μείγμα ενεργείας από αυτό που έχουμε σήμερα και ιδίως από το μείγμα προς το οποίο πορευόμαστε τώρα. Όλα αυτά έγιναν σε μια περιοχή όπου δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ανησυχία σε σχέση με την ασφάλεια τροφοδοσίας. Δεν είχε αντιμετωπιστεί καν τότε η πολιτική αντιμετώπιση της ε, κλιματικής αλλαγής. Ήταν βασικά μια ηλεκτροδότηση που βασιζόταν στον άνθρακα και το φυσικό αέριο, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και οι απεξαρτησμένες από τον άνθρακα τεχνολογίες είναι τεχνολογίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο σταθερό κόστος, πάγιο κόστος και μικρό μεταβλητό κόστος, αντίθετα από τις συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή το μήνυμα το οποίο δίνει η αγορά δεν είναι επαρκές για να εξασφαλίσει η, να εξασφαλιστεί η απόσβεση του παγίου κόστους. Από την έποψη αυτή, η πολιτική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει σχεδιαστεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ε, συνεκτικό, ακολουθώντας το μοντέλο που βασίζεται μονάχα στην ε, παραγωγή ενέργειας στα κράτη-μέλη και το μοντέλο της αγοράς δεν μπορεί να δώσει ένα μακροχρόνιο μήνυμα το οποίο μπορεί να προσελκύσει και να δώσει κίνητρα στις, στις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για μια ενεργειακή μετάβαση. Και επίσης δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ευκαμψία που χρειάζεται ένα σύστημα για να αντιμετωπίσει ανανεώσιμες ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση καταλήγουμε σε μια αγορά η οποία δεν λειτουργεί. Είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν δίδει κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων. Και όπως λέμε, μόνο οι χώρες οι οποίες έχουν ε, μεγαλύτερες ικανότητες, οι χώρες οι οποίες έχουν περισσότερα περιθώρια, αυτές μπορεί να λειτουργήσουν. Να λειτουργήσουν. Λειτουργεί γενικότερα η αγορά όμως σε πολύ βραχυπρόθεσμη βάση και υπάρχει μια τεράστια διακύμανση σε σχέση με το κειμενόμενο κόστος που οδηγεί σε μια πλήρη έλλειψη κινήτρων για επενδύσεις. Λοιπόν, η κρίση είναι σοβαρή στην ευρωπαϊκή αγορά και δεν θα λυθεί Εάν δεν περάσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, μια τέτοια πολιτική απαιτεί μια αγορά ενέργειας και μια αγορά ικανότητας παραγωγής με ένα επίπεδο εναρμόνισης ή έστω συνδυασμού πολύ ψηλότερο από τη σήμερα, με ένα δίκτυο διασυνδέσεων πολύ μεγαλύτερο από την δυναμική η οποία έχει ακολουθήσει τη λειτουργία του συστήματος τα τελευταία χρόνια και φυσικά ένα πολύ πιο σοβαρό ρόλο ε, της αγοράς και για τις εκπομπές που δεν έχει στείλει τα κατάλληλα μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα τα οποία θα διασφαλίσουν την επένδυση στην ενεργειακή, ε, στην ενεργειακή προσωρινή φάση αν θέλετε αλλαγής του τύπου παραγωγής είναι κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει και στην αποκέντρωση του ενεργειακού μοντέλου. <coughs> δηλαδή αναθεώρηση του συστήματος ε, ε, τιμολόγησης, επενδύσεις σε ευφυή e e συστήματα τα οποία να υπολογίζουν σωστά και να προϋπολογίζουν την ενεργή ζήτηση και επίσης και αλλαγή του προτύπου συνεισφοράς των παραγωγών καταναλωτών το επίπεδο των παγίων μορφών κόστους έτσι ώστε το πρότυπο αυτό το ευρωπαϊκό να μπορέσει να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι είστε επιχειρηματίας και εγώ ήμουν επιχειρηματίας αλλά ποτέ δεν είχα ακούσει κάποιο επιχειρηματία να δίνει μια τόσο έντονη παρουσίαση νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθείτε με την πολιτική. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι ο Κάρι Χιτάνεν, ο οποίος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Βάρτσιλα και της Ένωσης ε, Εργοστασίων Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Okay, no. Sorry. Mr. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Κυρίως σε μένα με ενδιαφέρει εδώ ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος και κάποια ευκαμψία. Θα σας μιλήσω και για τις εμπειρίες της εταιρείας Βάρτσιλα. Είμαστε ευρωπαϊκή εταιρεία, έχουμε ωστόσο εμπειρία από διάφορες αγορές του κόσμου. Σας έχω ετοιμάσει και ολίγες διαφάνειες. Εάν εξετάσουμε τώρα την εξέλιξη των συστημάτων ενέργειας, είναι καθαρό ότι βλέπουμε μεγάλη αλλαγή. Στο παρελθόν, η σταθμοί παραγωγής ενέργειας ήταν μεγάλοι και αργή στις ε, αντιδράσεις τους. Βέβαια και το φορτίο ήταν προβλέψιμο. Το εμπόριο ήταν πάντα βασισμένο σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις και δεν υπήρχε πολλή ενοποίηση μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών. Βέβαια από τότε έχουμε περάσει, έχουμε κάνει μεγάλο δρόμο και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που υπάρχουν και πολλές ενδιάμεσες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας, δηλαδή μεταξύ αυτών και η ενέργεια των ανεμογεννητριών και επομένως οι παραλλαγές είναι πάρα πολλές. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο του δυναμικού της παραγωγής πρέπει να αλλάξει. Έχει λιγότερες ώρες λειτουργίας και όταν λειτουργεί, λειτουργεί για συντομότερα χρονικά διαστήματα. Η δε τάση είναι προς πιο βραχυπρόθεσμες ε, ε, συμβάσεις εμπορίας της ε, ενέργειας. Και το Power Plant Portfolio, μάλιστα, το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των μετοχών των διαφόρων σταθμών ενέργειας, έχει αλλάξει πολύ. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραγωγικές ικανότητες και χρειάζεται εξισορρόπηση. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ευκαμψία ή ευελιξία. Παλαιότερα είχε καλός ένα σταθμός παραγωγής ενέργειας να χρειάζεται ώρες ή και μέρες μέχρι ότου φτάσει στην φουλ παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό τώρα πλέον δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται να μπούμε σε ένα σύστημα πια όπου χρειάζονται ίσως λίγα λεπτά για να πάρει μπρος ο σταθμός ενέργειας. Χρειαζόμαστε σταθμού ενέργειας που να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους ταχύτατα και σε πολύ υψηλό βαθμό. Για να ανταποκρίνονται δηλαδή στις αλλαγέ κατανάλωση. Αλλά και επίσης να μπορούν και να σταματούν την παραγωγή τους ταχύτατα. Για παράδειγμα, το σταμάτημα της παραγωγής ενέργεια είναι σημαντικό για να μπορούν να παρισχρήσουν περισσότερο είναι όσιμες στο σύστημα εφόσον αλλάζει ο καιρός και υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή από τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, άνεμο, ήλιο κλπ. Αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Εξάλλου είναι κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παραγωγής ενέργειας, είναι επίσης σημαντικό για τη μείωση των εκπομπών και βέβαια για την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. Μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα πού μπορούμε να βάλουμε αυτή την ευελιξία ή ευκαμψία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας για παράδειγμα είναι ένας. Επίσης οι διασυνδετές, οι interconnectors παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Επίσης η ανταπόκριση στην ζήτηση που σημαίνει ότι η παραγωγή προσαρμόζεται στην κατανάλωση και αυτό έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει. Η αποθήκευση δε εκεί παίζει ρόλο η αποθήκευση νερού για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά σε τουρμπίνες που, χρησιμοποιούν, που παράγουν ενέργεια και ούτω καθεξής σε ε, συσσωρευτές. Γενικά χρειάζεται συνεργασία όλων των πηγών ευελιξίας στην πράξη. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι για πολλά χρόνια που μας έρχονται η παραγωγή της ενέργειας θα εξακολουθήσει πάντως να είναι η πιο σημαντική πηγή ευκαμψίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της αγοράς, πρέπει να σημειώσει κανείς ότι ο σχεδιασμός της αγοράς τίνει να φτιάξει ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού για κάθε πηγή παραγωγής ενέργειας. Ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός συνέταξε μελέτη πέρσι σχετικά με το κόστος των διαφόρων πηγών ευκαμψίας και το συμπέρασμα πέρσι λοιπόν ήταν τη Διεθνούς Αρχής Ενέργειας ότι το κόστος των αγωγών ήταν το μικρότερο. Σήμερα βέβαια δεν δίνει η αγορά μηνύματα για επενδύσεις. Άρα, πώς, ποια μπορεί να είναι η λύση, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τις αναγκαίες επενδύσεις σε ευκαμψία. Αυτό το ερώτημα δεν απευθύνεται μονάχα στα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας. Υπάρχουν και πολλά άλλα συστήματα ενέργειας που χρησιμοποιούν και ανανεώσιμες ενέργειες και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Παράδειγμα, η ERCOT στις Ενωμένες Πολιτείες καλύπτει ολόκληρο το Τέξας και το Τέξας έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. 11.000 ΜΒ το περσινό χρόνο και μέχρι το 17 θα το έχουν διπλασιάσει. Και έχουν το ίδιο δίλημα. Η αγορά δηλαδή δεν δίνει μηνύματα ότι χρειάζονται επενδύσεις. Και αντιμετωπίζουν και σημεία εχμής. Και ο τοπικός ρυθμιστής έχει αναθέσει διάφορες μελέτες για να εξέβει την καλύτερη δυνατή λύση και το συμπέρασμά του ήταν ότι δεν θα προχωρήσει σε ένα μηχανισμό ρύθμισης των ικανοτήτων γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικά δαπανηρό για τους καταναλωτές. Απεφάσισαν λοιπόν εκεί στο Τέξας να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την αγορά της ενέργειας με τις βασικότερες βελτιώσεις να αναφέρονται στο ότι οι τιμές, οι χοντρικές τιμές της ενέργειας ανταποκρίνονται στο κόστος και να προσφέρουν βέβαια και αξία για εύκαμπτες ικανότητες παραγωγής. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τώρα είναι ότι έχουν περίπου 8 γιγαβάτ νέων έργων που βρίσκονται στον αγωγό ή που χρηματοδοτούνται ιδιωτικά, βασισμένα κυρίως στο αέριο. και έχουν και έργα ανταπόκριση στη ζήτηση, demand response. Αυτά είναι ενθαρρυντικά βέβαια σημάδια ότι η αγορά μπορεί να αποδώσει και να δώσει τα απαραίτητα σημάδια για επενδύσεις εφόσον βελτιωθεί ακόμα παραπάνω. Παρόμοιες ερωτήσεις συζητούνται και εδώ στην Ευρώπη. έχοντας υπόψη τις εμπειρίες άλλων χωρών, αλλά βέβαια και της ε, εταιρεία ERCOT, το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί ώστε όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά έχουν την ευθύνη για την εξισορρόπηση, balancing responsibility. Ο παραγωγός ενέργειας δηλαδή, εάν δεν μπορεί να παραγάγει τα όσα έχει υποσχεθεί και προκαλεί έλλειψη ισορροπίας, αυτός θα πρέπει να λάβει το κόστος αντί να το μετακυλήσει στους καταναλωτές. Σε μια βάση πλήρους ε, εξορρόπησης του κόστους. Αυτό σημαίνει πιο σύντομες συμβάσεις trading, πιο ε, ασταθείς τιμές, αλλά είναι απαραίτητη, απαραίτητες επαραίτητα αυτά τα σημάδια που δίνουν οι τιμές, τα μηνύματα που δίνουν οι τιμές για την ε, αύξηση της ευκαμψίας. Και αυτό είναι και η βάση του σχεδιασμού της αγοράς. Δεν έχει αρνητική επίπτωση στο συνολικό κόστος γιατί θα αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος. Το συμπέρασμα λοιπόν που βασίζεται σε αυτές τις εμπειρίες είναι ότι η αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αναπτυχθεί έτσι ώστε να λαμβάνει τα μηνύματα για επενδύσεις, για να εξασφαλίσει δηλαδή ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστική η παραγωγή του ρεύματο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ηλεκτρικού ρεύματο. Ευκαμψία είναι κάτι βεβαίω που ε, υποστηρίζει, βρίσκεται στη βάση τη επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Ευχαριστώ κύριε Γιετάνεν. Αυτή τη ο κύριος Στατιέντε είπε ότι είχε υπάρξει πολιτικός. Ήταν στο... στην κυβέρνηση του Φελίπε Γκονσάλες, πολύ παλιά. Και τώρα τον κύριο Σόμερ, ο οποίος είναι, ο, ε, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, RESCOP EU. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είστε όλοι υποθέτω πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τα θέματα της μετάβασης, είστε ομόλογοι κατά κάποιο τρόπο, λέγομαι Ζήγουα Τζόμα, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ομάδων και Συνεργατικών Ομάδων Πολιτών για τις Ανανεώσιμες Πηγές. Είμαι επίσης ε, και πρόεδρος της Ένωσης ε, Παραγωγών Νεολικής Ενέργειας με 6,5 περίπου χιλιάδες μέλη. Η μετάβαση στον τομέα της ε, ενέργειας μπορεί να ονομαστεί επίσης μετάβαση στην δημοκρατία και στην συμμετοχή των πολιτών. Να σας εξηγήσω καταρχάς τι είναι το Ρεσκόπ. Ε, συμπτυγμένα το είναι θα έλεγα συνεργατική ομάδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ασχολούμεθα με την παραγωγή, την ανάπτυξη, ε, την πώληση υλικού και την παροχή υπηρεσιών και την δημιουργία μικρών δικτύων. Δεν ασχολούμαστε, δεν είναι μόνο ε, ομάδες παραγωγών που συνεργάζονται αλλά γενικότερα πολίτες που ασχολούνται με το θέμα της ενεργειακής μετάβασης. Τα τελευταία τρία χρόνια είχα την χαρά να μελετήσω και να ταξιδέψω στην Ευρώπη και να συναντηθώ με τα ρέσκοπ που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Συναντήθηκα με τις εθνικές ομοσπονδίες και με τις ομάδες των παραγωγών. Υπάρχουν 2.500 ρέσκοπ σε όλη την Ευρώπη που συνεργάζονται και καθίστανται σιγά σιγά ένας ουσιαστικός οικονομικός εταίρος. Αν κοιτάξει κανείς αυτούς τους συνεταιρισμούς και αυτές τις ομάδες των πολιτών έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους. Όλες αυτές οι ομάδες ε, με τις οποίες συζήτησα ξεκίνησαν σαν, σαν πρωτοβουλίες πολιτών που συζήτησαν το θέμα αυτό στο σπίτι τους, στο σχολείο και ένιωσαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να ελέγξουν τις εξελίξεις. Υπήρχε κρίση αλλά δεν ήταν και δική τους ευθύνη για την κρίση αυτή, την οικονομική κρίση, τη χρηματοπιστωτική ενεργειακή κρίση και πάλι δεν μπορούσαν τίποτα και σε σχέση με τα τρόφιμα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Θέλησαν λοιπόν να πάρουν μέρος στη διαμόρφωση της αγοράς ενέργειας. Θέλησαν να γίνουν ε, οικονομικές οντότητες και να ελέγξουν την ενέργεια. Συνεργάστηκαν και είπαν ότι αν δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις και νέες οικονομικές μονάδες, πώς θα διαμορφωθούν οι ομάδες αυτές. Και συναντήθηκαν λοιπόν και κατέγραψαν τις 7 συνεργατικές αρχές που για πρώτη φορά διατυπώθηκαν το 1844 στη βιομηχανική επανάσταση όπου οι εργάτες, οι πολίτες ήσαν αντικείμενο ουσιαστικά εκμετάλλευσης και θέλησαν κάποιοι πολίτες να ελέγξουν τις εξελίξεις αυτές και την εξουσία της αγοράς. Κάποιες λοιπόν βασικές αρχές είναι η εθελοντική ελεύθερη συμμετοχή. Είπαμε ότι κάνουμε μια επιχειρηματική ομάδα η οποία δεν θα αποκλείει κανένα. Είναι μια ελεύθερη ομάδα, ο οποιοδήποτε θα είναι σε θέση να πάρει μέρος. Κατέγραψαν λοιπόν στον κανονισμό τους ότι ο οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεύτερον, δεν έχει σημασία πόσα χρήματα συνεισφέρει κανείς μέσω της επιχείρησής του. Αυτό που έχει σημασία είναι να οργανωθεί κανείς με βάση την αρχή ένας άνθρωπος μία ψήφος, δηλαδή δημοκρατική διακυβέρνηση. Και ε, η προσπάθεια δεν ήταν να αυξήσουν τις κιλοβατόρες ε, ή την επιστροφή των χρημάτων τους, θέλουν τα κέρδη να διοχετευτούν στις κοινότητες περισσότερο από ότι στην ίδια την εταιρεία. Πώς συμμετέχουν οι πολίτες λοιπόν, είτε το κάνουν αυτό συλλογικά σε ομάδες ρέσκοπ, είτε το κάνουν σε ε, ατομική βάση μέσω των μέσω που έχουν στη διάθεσή τους. Των, ε, αυτών των ε, συστημάτων. Γι' αυτό ένα από τα πράγματα τα οποία είδαμε μέσω αυτής της ε, συμμετοχικής διαχείρισης ότι εσείς που είσαστε εδώ θα καταβάλλετε το τίμημα για την μετα... μετάβαση στην ενέργεια ως καταναλωτές, ως φορολογούμενοι, ως χρήστες του δικτύου και ως αποταμιευτές. Όλες αυτές οι επενδύσεις λοιπόν θα γίνουν είτε από τράπεζες είτε από συνταξιδοτικά ταμεία, αλλά όλα αυτά είναι χρήματα των φορολογουμένων. Η φυσική πόροι όμως είναι κοινά αγαθά τα οποία ανήκουν σε όλους μας και θα πρέπει να περάσουμε στην ιδιωτικοποίηση. Δεν πρέπει αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν κέρδη, αλλά για το κοινό ενεργειακό σύστημα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα ηθικό δικαίωμα να εξασφαλίσουμε και μία θέση στην αγορά ενέργειας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με μία αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένωσης όπου ο πυρήνας της Ένωσης αυτής είναι ο ίδιος ο πολίτης. Ο πολίτης μπορεί να αναλάβει την διεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης και να συμμετάσχει πλήρως στην αγορά ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια αγορά ενέργειας όπου στην θέση των ε, δύο ή 2,5 χιλιάδων ε, ενεργειακών εταιριών που είναι με το δικό μας σχήμα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες εταιρείες. Όταν μιλάμε λοιπόν για πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες αντιμετωπίζονται κυρίως ως καταναλωτές. Για μας όμως είναι ενεργά εμπλεκόμενοι στην διαχείριση της ζήτησης. Οι πολίτες λοιπόν εμπλέκονται σε όλο το σύστημα παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι λοιπόν, μπορούν οι συνεταιριστικές οργανώσεις των πολιτών να λειτουργήσουν ως πηγή ενέργειας και μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τις εταιρείε της ε, πληροφορικής που θα συνεργαστούν μαζί τους και να κάνουν πιο ευφυές το σύστημα. Δεν είναι λοιπόν μονάχα <clears throat> καταναλωτές αλλά είναι ενεργοί παίκτες. Και κάτι ακόμα. Με τα δίκτυα Τα δίκτυα είχαν πάντα παραδοσιακά μία ε, μονοπωλιακή θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι οι πολίτες είτε μόνοι τους είτε μέσα από δημόσιους φορείς και συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του δικτύου ώστε να υπάρχει κοινό συμφέρον μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή. Τι λειτουργεί λοιπόν σε βάρος των πολιτών. Είναι η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία. Από τη στιγμή που αλλάζει η νομοθεσία και γίνεται γραφειοκρατικότερη, είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξουμε τους κανονισμούς που αφορούν μία ε, εταιρεία. Και είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα παρά όταν είναι δημοκρατικά και αποκεντρωμένα οργανωμένα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την πολυπλοκότητα και την γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει στις μικρές μονάδες να αναπτυχθούν και να αναλάβουν το βάρος της αγοράς. Όταν ξαναρχίσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδοτεί τις μεγάλες εταιρείες και να ε, υποστηρίζει τους πυρηνικούς σταθμούς, όπως το Hinkley Point, τότε δημιουργείται μια κατάσταση όπου δεν υποστηρίζεται η μετάβαση στα αποκεντρωμένα συστήματα, αλλά δίδεται βοήθεια στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Αυτό μειώνει τη δύναμη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν να πούμε και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω κατά λίγον είναι ότι αν θέλετε να προχωρήσετε, αν θέλετε να θέσετε στο προσκήνιο τους πολίτες, εμάς δηλαδή και εσάς, στην αγορά ενέργειας, ως σημαντικούς παίκτες θα πρέπει να τους ενθαρρύνετε και να παράγουν και να καταναλώνουν, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δημιουργήσετε ένα γήπεδο που δεν γέρνει στον τομέα της ενέργειας, να υπάρξει στη διαδικασία ε, διαγωνισμών για την ενέργεια και μια στη δημόσια πολιτική. Αυτό θέλει να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε να μιλήσουμε για την προσπέλαση των ανθρώπων στην ενέργεια, δεν μιλάμε μονάχα για την ισότητα ανταγωνισμού. Μιλάμε για να υπάρξουν οι διαφορετικοί κανονισμοί που θα εξασφαλίσουν ότι όλοι έχουν την ίδια πρόσβαση στην αγορά. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν αυτούς τους κανονισμούς ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά τα επόμενα 500 χρόνια στην αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Ζώμα. Περνάμε στο γύρο των ερωτήσεων. Δεν θα θέσω εγώ ερώτηση εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας αν και πρέπει να εκπροσωπήσω τον εισηγητή, αλλά με ακούσατε αρκετά. Θα ακούσω τον κύριο Νίκα. Ο κύριος Νίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. και οι τρεις παρουσιάσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και γι' αυτό να μου επιτρέψετε να θέσω κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες. Πολλοί θεωρούν ότι άνω του 30% της ανανεώσιμης ε, ενέργειας ε, ε, είναι επικίνδυνο. Ποσοστό άνω του 30% ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μίξ. Ποια είναι η γνώμη σας και κυρίως θέτω το ερώτημα στον κύριο Ατιένθα, ο οποίος ασχολήθηκε και με τεχνικά θέματα. Δεύτερον, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Ίσως βέβαια να μην υπάρχει θαυματουργή λύση, αλλά λέμε ότι η διασύνδεση δεν ξεπερνάει το 10%. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα 90% κάπου θα πρέπει να τα βρούμε και αυτά. Ε, δηλαδή εσείς προτείνετε να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο στο επίπεδο του 10%. Και τελευταία ερώτηση σχετικά με τις επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες. Αυτό λένε κάποιοι έχει, έχει δημιουργεί προβλήματα στις αγορές, στρεβλώνει τις αγορές και δημιουργεί ε, θέματα τιμών εξαγωγής ε, τύπου dumping και αυτό αφορά και την Ρουμανία, τη δική μου χώρα. Α, να ρωτήσω και για την αποθήκευση. Μιλάμε πολύ για αποθήκευση, αλλά είναι κάτι το πολύ μακροπρόθεσμο, κάτι το οποίο θα αναζητήσουμε ή θα επιδιώξουμε σε 30 χρόνια. Ο κύριος ε, Κατίνεν αναφέρθηκε στα θέματα της αποθήκευσης. Διαρωτώ με ποιες είναι οι πρόπτικες, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας. Γιατί από ό,τι ε, βλέπω εγώ η άντληση, η υδραυλική αυτή δεν επιτρέπει παρά μόνο ε, να συγκρατήσουμε το 50% της ενέργειας και το υπόλοιπο 50% θα χάνεται στην ε, ατμόσφαιρα και το ίδιο ισχύει και για άλλες ε, μεθόδους όπως οι συσσωρευτές πεπιεσμένου αέρα αλλά σε 50 χρόνια, σε 30 χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται άμεσα. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχω καταλάβει τίποτα πολύ καλά. Ε, τι γίνεται όταν δεν υπάρχει ας πούμε παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια τη νύχτα. Τότε τι θα πρέπει να γίνεται, θα παρεμβαίνουν οι ε, συμβατικές μορφές ενέργειας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε 50 ΜΒ ηλιακής ενέργειας ε, θα πρέπει να δημιουργούμε και 50 ΜΒ παραδοσιακής συμβατικής Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά είναι κάποιες ερωτήσεις τις οποίες ε, θέτουν πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Έχει σημασία νομίζω να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Ο κύριος Ρούμπιχ για το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε βράχυπρόθεσμα, μέσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να βάλουμε στις σωστές ράγες την πολιτική μας. Ακούστηκε το ερώτημα ιδιωτικές ή κρατικές. Ο ένας θέλει βεβαίως να κάνει επενδύσεις σε ένα μέρος και ο άλλος σε άλλο. Το γεγονό είναι ότι πρέπει να συνεργάζονται. Το πιο σημαντικό είναι να μπει το στοιχείο του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας. Σε διάφορα επίπεδα χρειαζόμαστε τον ανταγωνισμό. Ήδη ο ανταγωνισμός είναι καλά ε, κατεστημένος στα ορυκτά καύσιμα. Αρχίζει τώρα και μπαίνει και στις ε, ανανεώσιμες ενέργειες. Το πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχουν, διαφορετικό, υπάρχουν διαφορετικά κόστη. Δηλαδή όταν υπάρχει ηλιοφάνεια, όταν υπάρχει ε, βροχόπτωση που εξασφαλίζουν δηλαδή το νερό, από αυτά εξαρτάται ενώ στα ορυκτά καύσιμα εξαρτώμεθα από την ε, τιμή του πετρελαίου, από 150 δολάρια το βαρέλι στα 50, τα είδαμε τα πάντα πλέον. Είναι λοιπόν και το ερώτημα πώς μπορούμε ε, να συνδέσουμε τα μεγάλα συστήματα που είναι σημαντικά για τη βιομηχανία, ιδίω για την βιομηχανία Μεγάλη κατανάλωση ενέργεια, ένταση κατανάλωση ενέργεια, από την οποία ζει κυρίω η βιομηχανία στην Ευρώπη. Και το άλλο βέβαια είναι και οι οικονομίε κλίμακα. Και βέβαια, σημαντικό επίση, η ασφάλεια προμήθεια ενέργεια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μπορούμε να πετύχουμε μια εξισορρόπηση ανάμεσα στην ε, εξασφάλιση της προμήθειας ενέργειας από τη μια μεριά για τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις και από την άλλη μεριά οικονομίε οικονομίες που είναι σημαντική για τις μεγάλες βιομηχανίες. Και τελευταίο, έχουμε ένα πρόβλημα και με τις ε, προθεσμίες εγκρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε η Κομισιόν τελευταία, 11 χρόνια προθεσμίες για ε, ε, αδειοδοτήσεις. Το σχέδιο Juncker προβλέπει τώρα 3 χρόνια. Έχετε δει εσείς να υπάρχουν πραγματικά έργα μέσα στο σχέδιο Juncker που έργα που να μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε μια τριετία μαζί βεβαίως και με όλα τα συμπαρομαρτούντα, δηλαδή άδειε αδειοδότηση, χρήση, μάλλον αδειοδότηση, ε, χρήση, απόδοση και ούτω καθεξή. σα ευχαριστώ. Κύριο Σταμπουλάνο έχει το λόγο. Mr. Kelly. Ο κύριος Κέλλης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και τον συνάδελφο τον κύριο Ρουμπίκ θέλω να ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σα. Ετέθη το θέμα των επενδύσεων και της προσέλκυσης των επενδύσεων και της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης. Ο όλος στόχος του σχεδίου Juncker είναι ακριβώς η δημιουργία της εμπιστοσύνης, όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα, αλλά και σε όλους τους τομείς. Πιστεύετε ότι αυτά τα οποία έχουν προταθεί είναι εφικτά, πραγματοποιήσιμα Εάν όχι, τι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε το έφορο κλίμα όπου θα κινητοποιηθούν οι επενδυτές, ιδίως στην, ε, στο ενεργειακό τομέα και στις ανανεώσιμες κυρίως ενέργειες. Ο τελευταίος ομιλητής θα μίλησε για συνεταιριστικές ε, οργανώσεις παραγωγής, αιωλικές ε, ε μονάδες παραγωγής κτλ. Αυτό είναι ενδιαφέρον λοιπόν ως μια κίνηση εκ των κάτω προς τα άνω, γιατί δεν είναι ότι κάποιοι ηγέτες αποφασίζουν τι θα γίνει, αλλά είναι ο πληθυσμός απλώς ο οποίος το κάνει αυτό. Εγώ βρήκα στη δική μου εκλογική περιφέρεια στην Ιρλανδία μια αυξανόμενη αντιπάθεια, ιδίως κατά της ε, αιωλικής ενέργειας, είναι κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσμα έλλειψης πληροφορίας ή παραπληροφόρησης ή κάποιας τρομοκρατίας ή φοβίας που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τα αρνητικά αποτελέσματα των ολικών ε, γεννητριών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει πιστεύω να υπάρξει και περισσότερη κινητοποίηση αυτών των συνεταιριστικών οργανώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις και θα ήθελα να ζητήσω από τους ομιλητές να απαντήσουν πέντε λεφτά ο καθένας. Ο κύριος Ετιάνσα. Για την πρώτη ερώτηση, σχετικά με ποιο είναι το ανώτατο όριο στο οποίο μπορεί να καλύψει ε, ποσοστό ε, ε, εναλλακτικών μορφών. Δεν υπάρχει τέτοιο όριο. Εξαρτάται από το μίξ, εξαρτάται από το επίπεδο διασύνδεσης, εξαρτάται από το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Στην Ισπανία, στην παρούσα φάση, έχουμε ολική ενέργεια για 20% του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνουμε. Και κάποιες ώρες του χρόνου <clears throat> φτάνει και το 70% της στιγμιαίας κατανάλωσης ενέργειας. Έχουμε ένα ποσοστό εισχώρησης ε, των εναλλακτικών πηγών που μαζί με την ε, υδραυλική, υδροηλεκτρική φτάνει το 50 σχεδόν, πάνω το 40% εν Δεν υπάρχει μία απάντηση λοιπόν. Το θέμα είναι να διασφαλίσει κανείς ότι το σύστημα παρουσιάζει τις απαιτούμενες εγγυήσεις σε επίπεδο ικανότητας χρήσης του ηλεκτρικού διασυνδεδεμένου ευρύτερου συστήματος έτσι ώστε ε, για να αντισταθμίζονται οι ε, εναλλακτικές. 1450 ε, ΜΒ και θα φτάσουμε τα πάνω από 2.000 και θα φτάσουμε κάποτε και τις 10.000 με τα νέα δίκτυα. Γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή προωθούμε ένα, έναν εξαιρετικό συνδυασμό και με ε, backup την ευρωπαϊκή υπόλοιπη παραγωγή και έτσι μπορούμε λοιπόν να παρέχουμε την αντισταθμιστική ενέργεια όταν αυτή απαιτείται λόγω της πτώσης της παραγωγής εναλλακτικής. Λοιπόν, ε, μπορούμε να φτάσουμε στο 10% σε κάποιες βέσεις εναλλακτικής, είμαστε στο 3% τώρα. Εγώ είχα την δυνατότητα να, ε, να πάρω μέρος στην εκκίνηση εγκαταστάσεων που ασχολούνται με θέματα διασύζευξης είναι θέματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει και έχει παίξει πάρα πολύ θετικό ρόλο. Είναι η πρώτη τέτοια μορφή διασύζευξης ε, ήδη από το 1971. Δεν είχαμε φτιάξει τίποτα από τότε μέχρι σήμερα με τη γείτονά μας Γαλλία χρειάστηκε η πίεση της Ευρώπης, ε, μια συντονιστική ομάδα, η χρηματοδότηση και κυρίως η πολιτική όθηση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε όμως και πέραν αυτού. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις ικανότητες που έχουμε προώθησης κοινού ενδιαφέροντος προγραμμάτων. Έχω την αίσθηση ότι οι επιδοτήσεις και γενικότερα το σύστημα χρηματοδότησης των εναλλακτικών πηγών ε, ε, στρεβλώνει την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι προφανές αυτό οι ροές ανανεώσιμων ε, σε ορισμένες χώρες τεχνικά στρεβλώνουν τη συμπεριφορά του περιβάλλοντος συστήματος, αλλά σε οικονομικό επίπεδο ε, στην ουσία στρεβλώνουν και τις αντίστοιχες οικονομικές λειτουργίες των γειτονικών. Είναι όμως ε, μία μορφή ενέργειας, μία μορφή παραγωγής με ελάχιστες κειμενόμενες διαφοροποιήσει σε επίπεδο δαπανών και είναι προφανές και αναπόφευκτο ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εναρμονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο του συστήματος παραγωγής ανανεώσιμων. Τίθεται επίσης και το θέμα του με ποιο τρόπο θα οργανώσουμε τον ανταγωνισμό την Ευρώπη, πιο θεωρητικό. Η πολιτική αντιμετώπιση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών ασχολείται με θέματα παρεμβατισμού, δηλαδή ζητά ο πολίτης να μάθει ποιες είναι οι προτιμόμενες επιλογές στον τομέα της ενέργειας για λόγους αποδοτικότητας ενεργειακής, για λόγους καταποντέμησης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Το θέμα είναι πώς θα διαρθρώσει κανείς αυτές τις αλλαγές στην λειτουργία ορισμένων αγορών τις οποίες λειτουργεί ένα σύστημα που πρέπει όμως να γίνει πιο ε, αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η αγορά θα μπορέσει να δώσει κίνητρα σε επενδύσεις που θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί η ενέργεια και στον τομέα των εναλλακτικών πηγών και στον τομέα των δικτύων και πώς επίσης θα μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε το υπάρχον σύστημα με ένα ευφυή τρόπο και πώς επίσης θα μπορέσουμε να, να εναρμονίσουμε επαρκώς τους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν να λειτουργήσει το σύστημα ιδιαίτερα του ηλεκτρισμού με αυξημένα ποσοστά εναλλακτικών πηγών. Ανάλογα με τη ζήτηση και ανάλογα και με τη δυνατότητα παραγωγής καθυστέρησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, επόμενος Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρώτη ερώτηση. Αν δηλαδή 30% ανανεωσίμων είναι επικίνδυνο, αυτό που είδαμε είναι ότι όταν αυξάνει η συμμετοχή των ανανεωσίμων που είναι το όριο 20 με 30% είναι επίπεδο όπου το ποσόν πλέον των ε, ανανεώσιμων ενεργειών προκαλεί τεράστιες εναλλαγές και προκαλεί πρόβλημα στους υφιστάμενους παραγω... Ε, σταθμούς παραγωγής ενέργειας οι οποίοι δεν έχουν σχεδιαστεί να είναι ευέλικτοι. Αυτό είναι το δίλημα. Η ταχύτητα λοιπόν είναι ο βασιλιάς εδώ. Είναι ο κυρίαρχος. Όταν υπάρχει λοιπόν μέσα στο σύστημα ένα ποσοστό ανανεώσιμων, ποια μηνύματα δίνουν τότε στους επενδυτές να επενδύσουν σε ευκαμψία, σε ευελιξία. Αν δεν γίνουν οι επενδύσεις αυτές, τότε βέβαια υπάρχουν κίνδυνοι για το σύστημα. Αν γίνουν ωστόσο οι επενδύσεις, δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ο ρυθμός των επενδύσεων πάντοτε υπήρξε το πρόβλημα σε όλα τα συστήματα παραγωγής ενέργειας, διότι βέβαια ο σχεδιασμός βασίζεται στο παλιό σύστημα, όπου βάση για, το, για την επένδυση ήταν η μελέτη σκοπιμότητας του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Οι κιλοβατόρες που παίρνατε από το ε, σταθμό, αυτή ήταν, αν τώρα έχετε ένα τέτοιο ε, ευπροσάρμοστο σταθμό ενέργειας, δηλαδή μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα, αυτό είναι κέρδος. Αλλάζει λοιπόν το περιβάλλον. Δεύτερη ερώτηση τώρα που αφορά ιδιωτικό ή δημόσιο και ανταγωνισμό. Εγώ πάντως πιστεύω ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις μέσω του ανταγωνισμού, μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι επίσης σημαντικό οι πολιτικές να είναι συνεπείς και οι πολιτικές να παρεμβαίνουν στις αγορές όσο το δυνατόν, οι πολιτικοί μάλλον να παρεμβαίνουν στις όσο το δυνατόν λιγότερο Εφόσον υπάρχει επένδυση που βασίζεται στις αναμενόμενες τιμές, αυτό είναι καλό. Γιατί καλύπτει τότε κάποιο κενό μέσα στο σύστημα, κάποια ανάγκη του συστήματος. Και μέσω της επένδυσης αυτής, της ιδιωτικής επένδυσης, βελτιώνεται η συνολική ευελιξία του συστήματος και έτσι το όλο σύστημα αποδίδει καλύτερα. Είναι γεγονός ότι για πολλούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας αλλάζει τώρα το περιβάλλον και είναι σημαντικό στις μελλοντικές αποφάσεις να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τα αποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις, να μπορούν δηλαδή να αποκρίνονται με ταχύτητα. Αυτό διευκολύνει. Τελευταία ερώτηση σας τώρα. Αν θα είναι αποδοτικό το σχέδιο Juncker. Βέβαια εγώ δεν είμαι ειδικό για αυτά τα πράγματα, αλλά κατανόησα ότι το σχέδιο Juncker βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις συνολικές επενδύσεις και επομένως ίσως βέβαια το, το σχέδιο Juncker μόνο του να μην αρκεί για να λύσει το πρόβλημα. Αν όμως υποστηρίξει την, το σχεδιασμό της αγοράς, αν δηλαδή υπάρχει ευκαιρία για τον ιδιώτη επενδυτή να επενδύσει τα χρήματά του και να αποκομίσει κέρδος, τότε αυτό θα είναι θετικό. Ευχαριστώ κύριε Γιετάνεν Α, κύριε Ζόμερ Κύριο Σόμερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κέλλη έθεσε ένα ερώτημα σε μένα ειδικά μιλήσαμε για την τεχνολογική μετάβαση, αλλά ο Σκέλη Κέλλη τόνισε το πιο σημαντικό θέμα της μετάβασης που είναι η κοινωνική αποδοχή των ε, τρόπων παραγωγής ενέργειας. Βλέπουμε μεγάλη αντίδραση σε πολλές χώρες για τις ε, αιωλικές γεννήτριες, αλλά στην Ολλανδία ο Ολλανδός ε, έχει μία Ε, στάση που οδηγεί την κυβέρνηση στο να μην χρησιμοποιούν εγχώριους πόρους αλλά φέρουν καναδικό ξύλο για να το καίνε στα τσάκια τους. Οι πολίτες λοιπόν δεν δέχονται την μετάβαση στον τομέα της ενέργειας. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Και εφόσον δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτες θα αποτύχει η ενεργειακή μετάβαση. Μπορείτε να χτίσουν καλύτερες τεχνικές στην καλύτερη πληροφορική. Αλλά αν οι πολίτες πούν δεν θα πληρώσουμε πια για την ενεργειακή μετάβαση, πάπαλα η μετάβαση. Δεν πρόκειται να συνεχίσει. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις για την ενεργειακή τροφοδεσία. Μπορούμε να τις δημιουργήσουμε αυτές. Η λογική όχι στη δική μου περιοχή. Αυτό δεν αφορά τις ανανεώσιμες ενέργειες. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Έχει αλλάξει το περιφάλλον με τις αιωλικές. Βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι τις βλέπουν αυτές οι γεννήτριες αλλά δεν παίρνουν τίποτα από αυτές. Πηγαίνουν μακριά τα κέρδη από την τοπική οικονομία. Και γι' αυτό οι άνθρωποι είναι εναντίον, γιατί λένε αυτό δεν είναι δίκαιο. σε το περιβάλλον μου, βάζετε μια τουρμπίνα μπροστά στη μύτη μου, αλλά εγώ δεν παίρνω καμία προσθέμενη αξία, ούτε εγώ ούτε η τοπική κοινότητα. Όταν τώρα πάμε σε μια κοινότητα και πούμε τους λέμε να συμμετάσχετε. Και θα πάτε κι εσείς έσοδα από την αιωλική αυτή, από την αυτή εγκατάσταση αυτή. Θα πάρει η τοπική κοινότητα και έτσι θα δημιουργήσετε βιώσιμη ανάπτυξη, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετική αυτή η συζήτηση που έχετε με τους πολίτες οι οποίοι δεν συμφωνούσαν μέχρι τώρα. Μπορείτε έτσι να τους κάνετε να δεχτούν την ενεργειακή μετάβαση και να καταλάβουν γιατί είναι απαραίτητη η ενεργειακή μετάβαση. Χρειάζεται λοιπόν εκ των κάτω προς τα άνω δημοκρατικά να γίνει αυτή η οργάνωση για τα ενεργειακά θέματα. Δεν είναι μοναχα πρωτοβουλίε, δεν είναι ενώσεις καταναλωτών. Μιλάμε για εταιρείε οι οποίες θα κυριαρχήσουν στην ενεργειακή αγορά αν τους επιτρέψετε να λειτουργήσουν σε μια σωστή εσωτερική αγορά ενέργειας και για τις επενδύσεις. Κάποιος ε, ανησυχούσε για τις επενδύσεις που χρειάζονται. Στις κάτω χώρες έχουμε 350 εκατο, ε, δισεκατομμύρια αποταμίευσης. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα αιωλικό πάρκο στην Νότια Ολλανδία με μια μικρή συνεταιριστική οργάνωση η οποία θέλει να την υποστηρίξει 120 μέλη τα οποία θα γίνουν 200 μέσα σε μία εβδομάδα είχαν μαζέψει το απαραίτητο κεφάλαιο για αυτήν την αιωλική εγκατάσταση και ιδίω με χαμηλές με χαμηλά τραπεζικά επιτόκια υπάρχουν οι αποταμιεύσει, υπάρχουν τα λεφτά και μπορούμε να τα συλλέξουμε αυτά τα χρήματα και να τα επενδύσουμε. Εάν πείσετε αυτούς τους πολίτες να συμμετάσχουν και να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβαση. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά λοιπόν που ήθελα να πω. Δώστε στους πολίτες δυνατότητα να είναι ενεργοί, κάντε τους να χρηματοδοτήσουν ενεργειακή μετάβαση, δώστε τους τον έλεγχο των εσόδων, κάντε πιο δημοκρατικό το σύστημα, ώστε εμείς ως πολίτες μπορούμε να ελέγχουμε το δίκτυο και έτσι θα κάνουμε την ενεργειακή αγορά πιο ασφαλή για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σόμερ. Και τώρα είναι η ευκαιρία να δώσουμε στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Βέστροπ το λόγο. Έχετε πέντε λεφτά κύριε Βέστροπ για να απαντήσετε σε όλα αυτά τα οποία ακούσατε σήμερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο, όπως επίσης και τους εκπροσώπους ε, των εμπλεκομένων κατηγοριών επαγγελματιών που έχετε προσκαλέσει σήμερα. Το θέμα το οποίο σας απασχολεί είναι μία από τις πέντε διαστάσεις του συνολικού προγράμματος των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από την αποδοτικότητα στην ενέργεια και θα αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο μέλλον. Ήδη σήμερα αναφερθήκαμε στη σύνδεση ανάμεσα στην προμήθεια, στην διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας και στην κατανάλωση ενέργειας είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στην παρούσα φάση στο στάδιο της προετοιμασίας συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Έχουμε 15 σημεία δράσης, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα της πρωτοβουλίας. Νομίζουμε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα καλύψουν στο μέλλον τους στόχους τους οποίους έχουμε στον τομέα της ενέργειας. Πολλά από αυτά έχουν σχέση με αυτά που συζητήθηκαν σήμερα. Θα είμαι σύντομος, αλλά θα αναφερθώ όμως και στην πιο σημαντική από τις πρωτοβουλίες αυτές, την αγορά ενέργειας. Είναι μια βασική πλευρά των στόχων που έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Και ο Επίτροπος Καλνιέται έχει επίσης ε, αναφερθεί στο θέμα αυτό και έχει πει ότι πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα υπάρξει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρξουν περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην προπαρασκευή όλων μας. Αυτό θα ακολουθηθεί από την πρωτοβουλία του 2016 που θα φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας Ένα από τα θέματα που μας απασχολεί είναι το πώς σαν παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τα θέματα συμπαραγωγής τα οποία υπάρχουν σε διάφορες χώρες και πώς αυτό θα γίνει χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια στην αγορά ενέργειας. Ένας άλλος τομέας παρέμβασης είναι το πώς οι μελλοντικές αγορές ενέργειας θα είναι κατάλληλες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές. Από την άλλη θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και για την προετοιμασία της εφαρμογής των μέτρων για το 10% στον τομέα της, ηλεκτρικής, της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πώς θα φτάσουμε επίσης και στον στόχο του 15% που θα συμφωνήθηκε που συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών στα πλαίσια της προοπτικής 2020. Τώρα για το φυσικό αέριο είναι ένας τομέας που θα μας απασχολήσει επίσης. Περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση. Αυτό είναι ένας βασικός στόχος στην αγορά του φυσικού αερίου και τέθηκε το θέμα και από τον τέος Πρωθυπουργό της Λιθουανίας περιφερειακή συνεργασία προκαλεί πάρα πολύ ενδιαφέρον από πλευρά των κρατών μελών. Είχαμε πολλές συζητήσεις πριν λίγες εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, για μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και περιμένουμε και εμείς ε, να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέσο. Αντικαθιστώντας τον εισηγητή μπορώ να κλείσω αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Κουμπίλιος έδειξε πως μια χώρα μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από ένα μονοπωλιακό προμηθευτή, το έκανε, το είπε με τρόπο πολύ σαφή, ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες μπορεί να λειτουργήσουν πολύ καλά, αλλά συγχρόνως τόνισε την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη Ευρώπη. Η κυρία Κέμφερτ μας έδωσε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων, δεν θέλω να αναφέρω όλα αυτά που είπε, και ζήτησε περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης ο κύριος Σαρτιέλθα με μια ιδιαίτερα συγκινησιακή ομιλία τόνισε τη σημασία του ηλεκτρισμού σε ό,τι αφορά τη μείωση της χρήσης άνθρακα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τόνισε την ανάγκη για αλλαγές σε τεχνολογικό επίπεδο και ρυθμιστικό επίπεδο επίσης και ζήτησε περισσότερη ολοκλήρωση των ενεργειακών πολιτικών στην Ευρώπη κ. Χιτάνεν τόνισε το ρόλο της εσωτερικής αγοράς και είπε ότι εδώ έχουμε το βασικό πυλώνα για μια πραγματική ενεργειακή ένωση και υπογράμμισε το ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία και μας έδειξε τρόπους για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτή τη μεγαλύτερη ευελιξία. Ο κύριος Σόμερ ε, μας είπε ποιος είναι ο εφάνταστος και δημιουργικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να περάσουμε από την ενεργειακή μετάβαση στην ενεργειακή δημοκρατία και επίσης υπογράμμισε την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή αυτών τα οποία πράττουμε και τόνισε την σημασία τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κύριο Βέστροπ αναφέρθηκε μερικά από τα 15 σημεία δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλου του ομιλητέ εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας, της ΙΤΡΕ. Υπάρχει τώρα κάτι στα διάφορα. Όχι. Η επόμενη συνεδρίασή μας με την προεδρία του κυρίου Μπούζεκ θα είναι στις 6 Μαΐου από τις 9 στις 12 και από τις 15 18 και 30 και από τις 12 ως τις 10, ε, από τις 9 μάλλον μέχρι τις 10.30 και 15-18.30 στις 7 Μαΐου τέρμα της συνεδρίας. ευχαριστώ.